Καμάλ θα αντικαθιστούσε τον ε, κύριο Καρίμ για την παρουσίαση την έκθεση ε, για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία. Θα πιστοχωρήσουμε λοιπόν λίγο στην σε διάταξη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμάλ για τέσσερα λεπτά και μετά θα ακούσουμε τον Επίτροπο Μισελ. Θα γίνει η παρουσίαση λοιπόν τη έκθεση ε, Ζαγιάτ Καρίμ για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι Καρίμ, τι Κεμάλ. Νομίζω ότι είναι κανονικό να φαντάζεται κανεί ότι υπάρχει μια σύγχυση. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω σε όλους τους παρόντες ότι είμαι ο Καμάλ και όχι ο Καρίμ. Επομένω, πολλοί μπερδεύονται εδώ πέρα που ακούνε τον Καμάλ αντί για τον Καρίμ και τον Καρίμ αντί για τον Καμάλ. Ο συνάδελφό μου πάντω ζητά συγγνώμη γιατί λόγω ασταθμήτων συγκυριών δεν μπορεί να είναι παρόν εδώ. Η έκθεσή του καλύπτει το εμπόριο στα αγαθά, στις υπηρεσίες, στην πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Και όλα αυτά τα οποία μπορούν να προχωρήσουν επί τη βάση του κοινού ψηφίσματος μεταξύ του ΕΛΚ και της ομάδας των φιλελευθέρων. Θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση η οποία εξα, εξαιρεί τον προστατευτισμό. Τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αναπτύξουμε τους δεσμούς μας με τον, εταίρο, με τον εταίρο μας αυτό που είναι η Ινδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις το 2007 για τη λεγόμενη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και μια προτιμησιακή συμφωνία, όπως θα λέγανε ορισμένοι. Ο στόχος είναι μια ισορροπημένη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας που θα αυξήσει την πρόσβαση στις αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε πολλές περιοχές περιλαμβάνοντας και ορισμένα στοιχεία για την διαφάνεια των ρυθμίσεων σε τομείς επενδύσεων και υγειονομικά και φυτο υγειονομικά μέτρα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διευκόλυνση του εμπορίου και του τελωριακού καθεστώτος. Το κύριο σημείο της έκθεσης είναι το εξής, ότι αν εξετάσουμε το εμπόριο στις, στα αγαθά, έχουν μειωθεί οι δασμοί και είναι πλέον συγκρίσιμοι με αυτούς που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ασίας. Είναι περίπου 14% κατά μέσο όρο, ενώ είναι 4,5% γενικά οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Ινδία ανησυχεί για τις συνέπειες του προγράμματος REACH, και της, ε, του κόστου συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής αγοράς. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Τονίζει επίσης ότι η έκθεση ότι δεν θα πρέπει να θυγούν υπηρεσίε δημοσίου χαρακτήρα. Θα πρέπει να τύχει αναγνώριση το γεγονό ότι πολλέ φορέ το κράτο δεν είναι σε θέση να δώσει τι λεγόμενε δημόσιε υπηρεσίε και επομένω υπάρχει και ένα ρόλο για τον ιδιωτικό τομέα, για μη κρατικού φορεί οι οποίοι παρέχουν βασικέ υπηρεσίε στου φτωχού ιδίω όταν το κράτο το ίδιο δεν μπορεί να το πράξει λόγω ελήψεως εσόδων. Οι εμπορικέ ροέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ινδία είναι κάπω μη ισόρροπε. ενώ η Ινδία εξάγει περίπου το 9% του ΑΕΠ τη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη εξάγει μονάχα το 1,5%. Στο εμπόριο πάντως υπηρεσιών θα μπορούμε να έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στην ικανότητα των ειδικών εταιριών να αντιμετωπίσουν μεγάλες ροές δεδομένων και εδώ υπάρχει η ανησυχία για την προστασία των δεδομένων. Επίσης αναγνωρίζει η έκθεση ότι τα θέματα της επένδυσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί με, την κατάλληλη, τους κατάλληλους ε, τρόπους και δεν θέλουμε η Κομισιόν να έχει ελέγχους κεφαλαίων και εμπόδια στις κεφαλαιοικές ροές, ιδίως για τις φτωχές χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Επίσης τονίζει η έκθεση την προσήλωση της Τουρκίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και την ε, χρήση της σύμβασης TRIPS για την πνευματική ιδιοκτησία. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι οι υπερβολικές ε, ε, πιέσεις για τη δημόσια υγεία μπορεί να οδηγήσουν και σε μη προσβασιμότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους φτωχούς γιατί δεν μπορούν οι εταιρείε να αναπτύξουν φτηνά φάρμακα για αυτούς τους πολίτες. Επίσης η έκθεση αυτή αναγνωρίζει ότι ένα κεφάλαιο ανάπτυξη είναι βασικό στοιχείο οποιασδήποτε εμπορική συμφωνία και θα πρέπει να αναπτύξουμε το εμπόριο και τι επενδύσει, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την υγεία των εργαζομένων, τα πρότυπα στον τομέα του περιβάλλοντο και θα πρέπει συγχρόνω να γνωρίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να βρούμε κάποια ισορροπία μεταξύ των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος, των στάντα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και των αναπτυξιακών θεμάτων. Πολλές φορές η πλάστικα πηγαίνει στο ένα άκρο και δίνουμε υπερβολική σημασία σε μία πλευρά και ουσιαστικά καταδικάζουμε τις φτωχές χώρες σε περισσότερη ένδια γιατί δυσκολεύουμε το να μπορέσουν να αναπτύξουν παραγωγική ικανότητα οι εταιρείε στις φτωχές αυτές χώρες. Ευχαριστώ. Ο κ. Μισελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον που έδειξε για την κατάρτιση μιας συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ινδίας και να ευχαριστήσω και τον κύριο Καμάλ και την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου που κατήρτισε την έκθεση αυτή. Ε, καθώς επίσης και τις άλλες επιτροπές που ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία. Έγινε μια πολύ διεξοδική συζήτηση στο Κοινοβούλιο, καλύφθηκαν όλες οι πτυχές της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ινδίας που θα αποτελέσει τη βάση για την πιο πλήρη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γενικό πλέξιο και το περίπλοκο χαρακτήρα των σχέσεών μας με την Ινδία για να αναφέρω μόνο μία βασική πρωτοβουλία την οποία να επιζητούμε με την Ινδία και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και να συνάψουμε ε, μία συμφωνία ελευθέρου, των αναργών με την Ινδία προς όφελος και των δύο πλευρών ε, και αυτός είναι ο βασικός στόχος μας κατόπιν της μελέτης η οποία έγινε από ανεξάρτητο μελετητή και ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να αναλύσει το περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό πλαίσιο των επιπτώσεων και η αηφόρος ε, ανάπτυξη εξετάζεται για να μπορέσει και αυτή να καλυφθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να σας πω που βρίσκονται αυτές οι διαπραγματεύσεις οι οποίες ξεκίνησαν από το 2007 η τελευταία συνεδρίαση ήταν 17 με 19 Μαρτίου στο Νέο Δελχή, Μαρτίου στο Νέο Δελχή και προβλέπουμε να έχουμε ολοκληρώσει πριν από την διάσκεψη κορυφής. Ε, παρόλο που χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά ακόμη, είχαμε καλές συζητήσεις σε ορισμένους τομείς των υπηρεσιών και συζητήσαμε το κείμενο σε όλους τους τομείς της συμφωνίας, αλλά πριν ε, ολοκληρώσω θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Επιτροπής προς τον εισηγητή και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη. Σας ζητώ συγγνώμη κυρία Μπατζελή. Φτάσαμε επιτέλους και στη δική σας έκθεση με θέμα τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές στην επιτροπή γεωργίας αλλά και τις τέσσερις συναρμόδιες επιτροπές της επιτροπής